πρώτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας παρακαλέσω να σηκωθείτε για τον ύμνο της Ευρώπης. Liebe Kolleginnen und Kollegen. και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ε, καλωσορίζω εγκάρδια στην ε, πρώτη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις ε, εκλογές. Συγχαίρω όσους επανεξελέγησαν και όσους εξελέγησαν για πρώτη φορά. Κάτι λιγότερο από τους μισούς 700, από τους 736 βουλευτές εξελέγησαν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα ικανοποιητικό είναι το ότι 35% των βουλευτών είναι γυναίκες, το υψηλότερο ποσοστό μέχρι σήμερα. «170 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν στις εκλογές και η